Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ε, συνεχίζουμε. Ε, α, το λόγο έχει η κυρία Ποδηματά, παρακαλώ. Άννη. Thank you very much, President. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ως συνυπογράφουσα του ψηφίσματος για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, και εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας που πρέπει να προλάβει μία πτήση θα ήθελα να σας ζητήσω αν συμφωνήσει ε, εδώ ε, το τμήμα να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη και να ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα μετά το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης για τις ε, γενικευμένες δεσμολογικές προτεμήσεις. Είναι έκτακτη το το αίτημα αυτό, αλλά έχουμε έκτακτες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει κανείς διαφωνία, η κυρία Γιαννάκου. Παρακαλώ, κυρία Γιαννάκου. Κύριε Πρόεδρε, έχει δίκιο κυρία Ποδηματά για τους ίδιους λόγους που εξήγησε και εγώ με τη σειρά μου. Ζητώ το ίδιο. Δηλαδή, πριν ε, από το ψήφισμα να περάσουμε στην ψηφορία για τα φορολογικά θέματα. Ευχαριστώ. Διαφωνεί κανείς με την πρόταση αυτή. Αν όχι, αλλάζει η σειρά της ψηφοφορίας όπως προτάθηκε. Ο κύριος Οντή. Oui, Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να διαφωνήσω με την πρόταση αλλά επειδή κάθονται οι συνάδελφοι σιγά σιγά και οι πολιτικές ομάδες ετοιμάζονται να είστε σας παρακαλώ ε, πάρα πολύ συγκεκριμένος να μην πηγαίνετε γρήγορα έχουμε μια σειρά στις ψηφοφορίες συγκεκριμένη λάθη έχουν γίνει κατά το παρελθόν γι' αυτό σας παρακαλώ να μην τρέχετε πολύ Μην ανησυχείτε κύριε Οντή σημειώνουμε και δεχόμεθα την πρόταση της κυρίας Ποδηματά και της κυρίας Γιαννάκου και θα σας το πω ε, με τη σειρά. Πρέπει να σας κάνω μια ανακοίνωση. Ο κύριος Βλάντιμιρ Ρέμεκ με ενημέρωσε ότι παρετείται από μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 16 Δεκεμβρίου 2013 και με ενημέρωσε σχετικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού, διαπιστώνει τη χειρία της έδρας από τις